Καλημέρα παρακαλώ, καθίστε. inserire la vostra carta Να βάλετε και την ε, κάρτα ψηφοφορία στην ε, ισοχή του μηχανήματο σα. E και θα προχωρήσουμε στην πρώτη ψηφοφορία, δοκιμή, τεστ. Παρακαλώ λοιπόν να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Βάλτε τις κάρτες μέσα. Η δική σου είναι ανάποδα, τη βλέπω από εδώ. Με Φεράρι. όλα κάρτα, ο υπόστο, όλα μάνο. Λοιπόν, η κάρτα το μηχάνημα το χέρι, κάτι τρέχει. No. You can change seat. Μπορείτε να αλλάξετε θέση. Okay? Everybody's happy. Είμαστε όλοι ικανοποιημένοι. Είμαστε πολύ σκόρπιοι, είσαστε σκόρπιοι και είναι δύσκολα. Δύσκολη, δύσκολη αίθουσα αυτή. Let me see if something different. Mm. Okay, I will try.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 Okay. Il punto 10 all'ordine del giorno. Το σημείο 10 της ημερήσιας διάταξης προβλέπει ψηφοφορία. Σύσταση για δεύτερη ανάγνωση για κοινού κανόνες για τις διεθνείς οδικές μεταφορές εμπορευμάτων. Αναδιατυπωμένη εκδόση, Εισηγητή Ματιέ Κρόπς. Ψηφίζουμε τη συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. μπορούμε να ψηφίσουμε όλες τις συμβαστικές μαζί. Κοιτάξτε, έχω μια πρόταση, συμπληρωματική πρόταση. Να ψηφίσουμε σε δύο ομάδες ομάδα 1 συστάσεις του εισηγητού, δεύτερη ομάδα τροπολογιών, όλα τα υπόλοιπα. Να έχουμε δύο ψηφοφορίες σε κάθε μία. Πρόεδρος. Βήμα-βήμα. Αγάλι-αγάλι. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε τη συμβαστική, την ομάδα των συμβαστικών προτάσεων, ναι. Ψηφίζουμε λοιπόν συμβαστικές λύσεις υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται μέχρι τη συμβαστική υπαριθμών 11. Αυτό σημαίνει ότι έχουν εγκριθεί τροπολογίες μέχρι την 11 και τα άρθρα. Οι τροπολογίες 17 Πάμε στην τροπολογία 19. Στέρξ, Ένις και Πλασάρτ. Πρέπει να ψηφίσουμε την 17 και 28. Ήταν εντός της ομάδας, λέει ο Πρόεδρος. Ήταν εντός της ομάδας μετά την 29. Και όταν ξεκινήσουμε τη δεύτερη συστάδα τροπολογιών, τότε θα δούμε. Τροπολογία 19. Στέρξ, Βασκάρ λοιπά, Πλεσάρ. Ποιο είναι υπέρ. Στέρξ, Ένι, Πλασάρτ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 20 αποσύρεται. 20 22. Στέρξ, Ένι, Πλασάρτ. Υπέρ. κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 23. Βόλτμαν Κόλ, Δεγκάντ Πασκουάλ, Ζαβερμπόφσκι. Υπέρ. Κατά. Αποχέ. Απορρίπτεται. 24 Χαρντίμ Αποσύρω την 24. Καλώς. Αποσύρω την 24 λέει ο πρόεδρος. Πάμε. Στην τροπολογία 25 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται οι άλλες αποσύρονται πάμε στην τελική ψηφοφορία ψηφίζουμε λοιπόν τη σύσταση που τροποποιήθηκε υπέρ μάλλον ξεκινάμε την ψηφοφορία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 34 παρόντες, 33 ψηφίσαντες, 25 υπέρ, 6 κατά, 2 αποχές εγκρίνεται. Ωραία. Συγχαρητήρια θα τα δώσουμε στον κύριο μετά την άλλη ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τη δεύτερη έκθεση κοινοί κανόνες για πρόσβαση σε διεθνείς αγορές για πούλμαν και λεωφορεία. Πρόσβαση στην αγορά των μεταφορικών υπηρεσιών με πούλμαν και λεωφορεία. Ψηφίζουμε όλες τις συμβαστικές προτάσεις μαζί. Συμφωνείτε? Μάλιστα. Ψηφίζουμε συμβαστικές τροπολογίες από την 1 μέχρι την 8 υπέρ κατά αποχές οι συμβαστικές εγκρίνονται. Συμπεριλαμβαναμένης τις 11 και 8. Όλη η γκρίζα ζώνη καλύπτεται. Τροπολογία 12. Βόρτμαν Κόλ και Τικάου έχουν αποσυρθεί και η 14 κατέπεσε. Άρα τελική ψηφοφορία. Τελική ψηφοφορία. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 34 ψηφίσατε, 32 υπέρ, 0 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται, συγχαρητήρια στον κέντρο Ψηφίζουμε το άλλο πακέτο για, τα, εξωτικές μεταφορές. Σύσταση σε δεύτερη ανάγνωση. Κυρίες ίσως όσον αφορά τις, τους όρους που πρέπει να πληρούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του οδικού μεταφορέα η η κυρία Σίλβα Αντριάννα Τσικάου. Και εδώ έχουμε τις συμβαστικές τροπολογίες, προτείνω, τις προτείνουμε να τις ψηφίσουμε όλες μαζί ομαδικά, ποιος είναι υπέρ των συμβαστικών, κατά, αποχές εγκρίνονται, όλες οι άλλες αποσύρονται και εδώ λοιπόν πάμε στην τελική ψηφοφορία που ξεκινάει.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 34 ψηφίσαντες, 34 υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην κυρία Τσικάου. Ωραία. Είμαι πολύ ικανοποιημένο. Πάει και ο δρόμος. Πάμε στο σημείο 13 της ημερήσιας διάταξης. Έκθεση Ντουσού. Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο για ανταγωνιστικέ εμπορευματικέ μεταφορέ. Είστε έτοιμοι. Ψηφίζουμε την τροπολογία 31. Λάιχτφριντ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 σαβαρή υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Προτείνω να ψηφίσουμε ομαδικά τις τροπολογίες 61, 63, 65, 66, 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται όλες. Εξήντα δύο, ορτουέντο λαρέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 Σίμψον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 Σίμψον τροπολογία 70 για Alexander υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 69 Σίμψον υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Εξήντα οχτώ ορτών υπέρ. Κατά. Θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Πέρας ψηφοφορίας. 19 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. Πάμε τώρα στην 71 Jacobs υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 72 Ταυτόσημη με την 63 Κράμερ υπέρ. Συγγνώμη, είναι με την 73 ταυτόσημη. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 74 Κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 75 Ορτουάντο Λαρέα υπέρ. Κατά. Αποχές θα γίνει ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ηλεκτρονικού ελέγχου. 19-14 εγκρίνεται ή 75. 76 που τη χαιρετίζουμε που έφτασε γέρο υπέρ κατά πρέπει να γίνει έλεγχος για την 76 για άλλα σέντερ ηλεκτρονικός έλεγχος Πέρας ψηφοφορίας. 17-17. Δεν εγκρίνεται. 8 του συγητού υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 Αλμπερτίνη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτουν οι 78 και 79. Πάμε στην 80 για Λασέντερ υπέρ. Πρέπει να ψηφίσουμε την 77 τελικά Αλμπερτίνη υπέρ. «78 ψηφίζουμε υπέρ» «Κατά» αποχές απορρίπτεται 79 σαβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 80 γέλα σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 γέλα σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρινέται 84 σαβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 του συγκητή υπέρ καταπίπτει μετά το 83 85 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 86 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 87 υπέρ κατά και έχει σβήσει το μικρόφωνο του Πρόεδρου δυστυχώς 88 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές 88 Μαρινέσκου υπέρ κάνουμε έλεγχο ξεκινάει ο έλεγχος Chiusa Πέρας. 17-17 δεν εγκρίνεται. Δεκαεφτά, δεκαεφτά δεν εγκρίνεται. Ογδόντα, Λάιτφριντ. υπέρ, κατά, Έλεγχος. Έλεγχος 89. 89. Έλεγχος. 14 20, υπέρ, 21 κατά. Απορρίπτεται. Σίμψον 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 αρτών δολαρέα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 94 για Αλεσάνδερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 92 Αλμπερτίν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 95 Σίμψον υπέρ αποσύρεται η 95 Σίμψον πάμε 96 και Καθώς είναι το 97, 100, 104, 112. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. Ένα 98 φουρέα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 καταπίπτει. 101 Γιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτω. An den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 Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 102. Τέλος. 19 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται η 102. And then Φίλε, Fino al 112 abbiamo Ήδη ψηφίσαμε αδικά μέχρι 112, είμαστε 113 κτλ. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 114 κρίμερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 115 ορτών δολαρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 116 τι υπέρ κατά αποχές απορρίπτει 117 σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ας γίνει η ηλεκτρονική επαλήθευση για την 117 σαβαρή ξεκινάμε για την 117 ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας 18 υπέρ, 18 κατά, δεν εγκρίνεται. Εκατόν δεκαοκτώ υπέρ. Κατά. Αποχές, ηλεκτρονικός έλεγχος και εδώ. Τέλος. 20-16 εγκρίνεται. 119 άλλα σέντερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100, απορρίπτεται συνέχεια, 120 χένι πλασάρ υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την 120 ένις πλασάρ. το όλοι. Τέλος 17 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. 121 για Λασέντερ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 122 Μαρινέσκου υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 123 Jacobs με την προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται 127. Ορτών δολαρέα με τη γνωστή προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 124. πίπτη, 125 Αλβερτίνη πίπτη και αυτή. 126 Σίμψον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 128 Λάχτφιντ υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται 129 Σίμψον υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 130 για Σέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 10 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 131 ορτών δολαρία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 132 κατά καταπίπτει. 11 του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 12 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 13 του υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 133 του υπέρ. κατά άποχες απορρίπτεται. Α, λέει ο πρόεδρο. 133 ορτουόντο λαρέα, όχι του συγητή. Έλεγχος για την 133 ορτουόντο λαρέα. Ψήφισα το λίγο. 37 ψήφισαν. Πέρας ψηφοφορίας. 21 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται το του εισηγητή για το τμήμα που δεν καλύπτεται από την τροπολογία 133. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Πάμε στην 134 ορτών δολαρέ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 135 Λάιχτριντ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 136 ορτουόντο λαρέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 ορτουόντο λαρέα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 thread, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 143 Hennis card, με προφορική τροπολογία που την ξέρετε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 139 ορτών δολαρία υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 140 φουρέ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 του εισηγητή πίπτη, Όπως και 141 142 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 144 τσικάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 145 μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 146 κρέμερ υπέρ. Κατά. Έλεγχος για την 146 κρέμερ. να πάρουμε και μια ανάσα. Πέρας επαλήθωσης. 15 υπέρ, 22 κατά, απορρίπτεται 148 Σίμψον υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 147 οτών δολαρέα υπέρ. Κατά. Θεωρώ ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε έλεγχο για την 147 ορτών δολαρέα. το όλοι. Ναι, πέρας. 20 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει 149 φορέ, πάμε 150 κρέμερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να κάνουμε έλεγχο για την Κρέμερ. Ναι, δεν σας κοίταζα. Ξεκινάει ο έλεγχος λοιπόν. Τέλος. 21 υπέρ, 16 κατά, Καμία αποχή. Εγκρίνεται η τροπολογία. 150. Κρίμα. 151. Jacobs υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 152. Simpson υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 153. Jacobs υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 του κατά καταπίπτει. 154 Kramer υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 155 Simpson υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 156 Μαρινέσκου. «156 Μαρινέσκου υπέρ» κατά αποχές απορρίπτεται. 17 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 157 Ένις πλασφάρ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος ψηφίσατε όλοι πέρασε 17 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 158 Simpson υπέρ, κατά, άποχες, επαλήθευση, έναρξης ψηφοφορίας. Πέρας. 18 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 159 σοβαρή υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 18 εισηγητή υπέρ κατά έλεγχος 18 του εισηγητή ψήφισατε όλοι πέρας 19 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται 160 Jacobs υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 19 του ηγητή υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται οπότε καταπίπτει 161 162 πάμε στην 163 ορτουόντα λαρέα υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος που ξεκινάει τώρα. Πέρας 18 υπέρ 19 κατά απορρίπτεται. Πάμε στην 163 του συγητή υπέρ. Α, συγγνώμη, 20. Υπέρ κατά αποχές η 20 εγκρίνεται. Συμβιβαστική 1 Σον Τζέικοπ, Ορτών Δολαρέα και Κρέιμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Οπότε καταπίπτει 166-165 μέχρι την 169. Καταπίπτουν όλες και ψηφίζουμε την 170 Κρέιμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 κάνει να καταπέσει 171 ορτών δολαρέα και ψηφίζουμε την 172 φουρέ βιράκ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική καταπίπτουν οι άλλες μέχρι την 193 και μετά 105 μέχρι 108 μένει 194 Light Street υπέρ καταπίπτουν μέχρι 193 και από 195 έως 198. Πρέπει να ψηφίσουμε την 194 Leichtfried. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται και αυτό. Πάμε στην 199. Ορτώντο Λαρέα και τη 200 Leichtfried. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτονται. 201. Jacobs υπέρ κατά δεν βλέπω χέρια μου φαίνεται ότι απορρίπτονται. Θέλετε να κάνουμε έλεγχο, ας κάνουμε. 201 Jacobs έλεγχος. Πέρας 15 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 26 της ηγητή υπέρ, κατά. Άλλος ένας έλεγχος για την 26 του ηγητή. Πέρας. 19 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική. Άρα καταπίπτουν 27, 28, 203, Καταπίπτουν όλες οι τροπολογίες μέχρι τη 214 σαβαρία που ψηφίζουμε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 215 Κρέμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 216 Κρέμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 217 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 218 Jacobs υπέρ κατά αποχές έλεγχος. 2.18 Jacobs έλεγχος. Πέρας. 15 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται 219 δισό υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται 220 δισό υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 221 ορτών δολαρία υπέρ, κατά έλεγχος 221 ορτούντο λαρέα πέρας 18 υπέρ 16 κατά εγκρίνεται 222 Jacob Zipper κατά έλεγχος 222. Jacobs. Πέρας. 19 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται. Καταπίπτει η 223. 224 φουρέ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 29. Πάμε στη 30 του συγκεκριμένου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.25 ορτών δολαρέα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται αλλά σε ελέγξουμε. Ξεκινάμε έλεγχο για τη 225. Ορτούντο. Ωραία. Τέλος. 18 υπέρ, 16 κατά, εγκρίνεται 226 κόστα υπέρ, κατά. Νομίζω ότι υπορρίπτεται 227 ορτών δολαρέα υπέρ. Όχι, να κάνουμε έλεγχο για 226. 226 κόστα. Έλεγχος. Ξεκινάει. Πέρας. Δίκιο έχετε. 15 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται. Λέει ο Πρόεδρος. Είμαι πολύ σεμνός. 227 ορτών δολαρέα. Υπέρ. Κατά. Αποχές από το 228 του σώμα υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 2.29 Σίμψον υπέρ κατά έλεγχος 2.29 Σίμψον πέρας 16 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται 230 Σίμψον υπέρ Νομίζω ότι είναι παρόμοιο. Θα το κάνουμε και αυτό, θα κάνουμε έλεγχο. Πέρας έλεγχο Όπως πριν 16 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται 2.31 κρέιμερ υπέρ. Κατά. Παιδιά, είμαστε πάνω στο, στη γραμμή πάντα. Πρέπει να κάνουμε έλεγχο για την Κρέιμερ. Τέλος ελέγχου. 15 υπέρ 19 κατά. Απορρίπτεται. 2.32 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 Κρέιμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 33 σοβαρή κατά αποχές εγκρίνεται 34 ορτών λαρέα είναι γλωσσική υφής πάμε στην τροπολογία του συγκητή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά θα κάνουμε παλήθευση. Τέλος. 19 υπέρ, 15 κατά, η 35 εγκρίνεται λοιπόν. Καταπίπτει 36 φουρέ. 37 σαβαρή τώρα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 Μαρινέσκου υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας γίνει επαλήθευση 38 Μαρινέσκου ηλεκτρονικός έλεγχος τέλος 21 υπέρ 13 ψήφοι κατά εγκρίνεται οι δύο του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η 39 σοβαρή και η 40 ορτούν δολαρέα. Πάμε στην 3 του συγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει η 41 ορτούν δολαρέα. Πάμε 42 ορτούν δολαρέα υπέρ. Κατά Έλεγχος 42. Ορτούντο Λαρέα. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψήφισατε όλοι. Τέλος. 18 υπέρ, 16 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. Η 42 ορτών λάρεα 43 σαβαρή υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι είναι όπως πριν αλλά είναι αδύνατο να διακρίνω. Ηλεκτρονικός έλεγχος, έλεγχος συγγνώμη, για τις 43 Σαβαρή. Τέλος. 16 ψήφοι υπέρ, 18 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. 4 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 44 ορτού αντολαρέα υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται 45 ορτών δολάρια έπερ κατά έλεγχος τη 45 ορτών δολαρέα ηλεκτρονικός έλεγχος μου φαίνεται ότι εγκρίνεται όμως ας κάνουμε τον έλεγχο ψηφίσατε όλοι Α, κάποιος δεν ψήφισε, εγώ ήμουνα, συγγνώμη. Τέλος ελέγχου. 18 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται 46 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Όπως πριν, εγκρίνεται. 47 Σαβαρή υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Να κάνουμε έλεγχο. Επαλήθευση λοιπόν. Τέλος. 16 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. 48 ένις πλασάρτ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 του εισηγητή υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 49 και υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάμε. Για τη 49 49ΔΕΒΕΙΡΑΚ ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 15 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. 50 σαβαροί υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά ας κάνουμε μια παλήθευση. Ορίστε. Τέλος ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται 51 ορτών δολαρέα υπέρ. Κατά. να κάνουμε έλεγχο έλεγχο. Να είναι καλά η ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 17 υπέρ, 16 κατά. Εγκρίνεται. 52 ορτών δολαρέα. με το 53 κρέμα υπέρ. Κατά αποχή απορρίπτεται 54 ενής πλασκάρτ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 55 κρέμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 δισόν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 57 σαβαρή υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος 57 σαβαρή ξεκινάμε Πέρας. 16 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. 6 του εισηγητή υπέρ. Είναι ταυτόσιμο με τα 58 ορτών δολαρέα. Λοιπόν, υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας κάνουμε επαλήθευσή όμως. Όχι. Δεν θέλεις επαλήθευση. Ας το υποστούμε και αυτό. Επαλήθευση για την 58. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Με μεγάλη πλειοψηφία εγκρίνεται. Ο Γιαζαμπόσκι δεν σφάλει ποτέ. 59 ορτών δολαρέα. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει επτά του εισηγητή, οπότε ψηφίζουμε την νομοθετική πρόταση αυτή όσα τροποποιήθηκε κοινά η ψηφοφορία. Τέλος, 34 ψήφισαν, 33 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Ψηφίζουμε το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. 32 υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στην κύριο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

Ευχαριστώ.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 Possiamo riprendere il posto. Συνεχίζουμε αγαπητοί συνάδελφοι. Don't worry. Be happy. Be ready. Be... Don't worry, be ready. Συνεχίζουμε τις ψηφοφορίες μας. Ψηφίζουμε για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές. Εισηγητής ο Μισελ Τεσενέ. Ψηφίζουμε την τροπολογία 43 του κυρίου Κύρκο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 44 Μπλόκλαντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 44 του κυρίου Μπλόκλαντ. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. 33 ψήφισαν, αλλά βλέπω μόνο 31. 19 υπέρ, 13 κατά. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η τροπολογία Blockland 44. Δεύτερη τροπολογία της, Επιτροπής, της Νομικής Επιτροπής υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 45, ναι. ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 46, Βόρτμαν Κόλ, υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 47 Μακάρθι, Χάρμπορ και ούτω καθεξής ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 48 Evans ποιος είναι υπέρ κατά ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 48 Evans άρχεται η ψηφοφορία τέλος ψήφισαν 20 υπέρ και 12 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 48 του κυρίου Evans. Τροπολογία 49, Στόκμαν. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 50. Μπλόκλαντ αποσύρεται. Τρίτη τροπολογία της Νομικής Επιτροπής. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 3 του εισηγητού είναι μια γλωσσική υφή. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. 51 τεσσένα. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία α. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχέ εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία α. Οπότε καταπίπτουν οι σχετικέ τροπολογίε με το άρθρο 3. Ποιο είναι υπέρ τη 5 τώρα, του εισηγητού. Τροπολογία 5, Ποιο είναι υπέρ. Ποιο είναι υπέρ τη 5 του εισηγητού. Κατά αποχέ εγκρίνεται 6 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ Τη τροπολογία 6. Κατά αποχέ εγκρίνεται 54 βλάστο. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 55 μπλόκλαντ υπέρ κατά αποχές μάλλον έχει εγκριθεί αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Τροπολογία 55 Blockland άρχεται η ψηφοφορία. Λήξη της ψηφοφορίας. Ψήφισαν 19 υπέρ και 14 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 55. Οπότε 56 του Βλάστο καταπίπτει. 57. Ποιος είναι υπέρ του κυρίου Evans της τροπολογίας 57. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 58. Κύρκοπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 59. Κύρκοπ. Υπέρ. Και 60. Ομού. Ποιος είναι υπέρ. 59 και 60. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 61. Κύρκοπ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 62. Κύρκοπ. Υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική τροπολογία Β. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται η συμβαστική τροπολογία Β. Τροπολογία 63 για Ζεμπόψκι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 64 με την προφορική τροπολογία Ζαρτίν Φερνάντες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον έχει απορριφθεί, αλλά καλύτερα να το ελέγξουμε. Τέλος της ε, ηλεκτρονικής επαλήθευσης. Ισοπαλία με 16 ψήφους και μία αποχή. Εγκρίνεται, εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. 7. Ποιος είναι υπέρ. τά του εισηγητού. Κατά αποχές εγκρίνεται. 8 του εισηγητού ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 9 του εισηγητού υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 65 Βόρτμαν Κόλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 66 Μπλόκλαντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 67 Κώστα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Α, ηλεκτρονικός έλεγχος για τροπολογία 67. Aware, but I had the coffee people, you know, that's in front of me. Luckily, because otherwise I would disappear. Thank you very much. Plenty of. Allora è provato. Α, ναι, δεν sorry. Α, sorry, sorry. Είπα, εγκρίνεται, αλλά ξέχασα να πραγματοποιήσω τον ηλεκτρονικό έλεγχο. Τέλο τη ηλεκτρονική ψηφοφορία, 18 υπέρ, 15 κατά, όντως εγκρίνεται. Η τροπολογία 68 του κυρίου Βλάστο ω ε, προσθήκη, ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές μάλλον έχει απορριφθεί 69 κόστα υπέρ κατά και αυτή μάλλον έχει απορριφθεί αλλά ας το ελέγξουμε όποιος φυλάει τα ρούχα του Chiuso. Τέλος της ψηφοφορίας, 14 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται η τροπολογία 69. Τροπολογία 10 του εισηγητού. Ποιο είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 70, Βόρτμαν Κόλ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 11 του εισηγητού, ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται 71 ναι. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 ναι. ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 το εισηγητού ποιος είναι υπέρ κατά Αβέβαια το αποτέλεσμα. Ας κάνουμε μια ηλεκτρονική επαλήθευση. Ψηφίσατε. Λήξη της ε, ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 16 κατά, χωρίς αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 12 του εισηγητού. 73. Μακάρθη και άλλων. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 74. Πισκόρσκι. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Όπως και πριν εγκρίνεται. Ψηφίζουμε σελίδιν της τροπολογίας 13 ως 1. 75, 14, 100, 101, 30, 31 και 1. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 76. Μακάρθη. Ποιος είναι υπέρ κατά, απορρίπτεται. Τέταρτη τροπολογία της Νομικής Επιτροπής, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 80, 82, 83 και 84 ομού, ποιος είναι υπέρ, κατά, Μια και είναι πολλές, ας κάνουμε έναν ηλεκτρονικό έλεγχο για καλό και για κακό. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε όποιον θέλετε, αλλά ψηφίστε. Τέλος του ηλεκτρονικού ελέγχου. 14 υπέρ, 18 κατά. Απορρίφθηκαν οι τροπολογίες. Τροπολογία 77 και 78. Grandes Πασκουάλ και Κίρκοπ παρόμοιες. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Απορρίπτονται. 79. Στόκμαν. Καλύπτεται, καλύπτεται. 81. Λίχτεμπεργκερ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον έχει εγκριθεί. Αλλά Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία, γιατί δεν σηκώνετε ευκρινώς τα χέρια σας. Λήξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, 18 υπέρ, 14 κατά. Εγκρίνεται η τροπολογία 81 της κυρίας Λίχτεμπέργκερ. Ψηφίζουμε τις τροπολογίες 15 και 85 που είναι ταυτόσιμες του εισηγητού και του κυρίου Γιαζαμπόφσκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 86 και 87 για Ζεμπόφσκι και Στόκμαν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Μάλλον έχουν απορριφθεί, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ηλεκτρονική επαλήθευση. Τέλος. 15 ψήφισαν υπέρ και 17 κατά. Χωρίς αποχές. Απορρίπτονται. Τροπολογία 16 του εισηγήτου ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 17 του εισηγήτου ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 88. Κύρκοπ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 89 Evans υπέρ. Κατά. Έχω την εντύπωση ότι εγκρίνεται, αλλά σε ελέγξουμε ηλεκτρονικά την τροπολογία 89 Evans. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος της ψηφοφορίας με 21 ψήφους υπέρ και 12 κατά έχει εγκριθεί 90 Evans, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 18 του εισηγητού καταπίπτει. και είχε αποσυρθεί η υπερπολογία 91. 92 Βλάστο, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 93 Blockland. Γλωσσική τροπολογία. Ψηφίζουμε ποιος είναι υπέρ της τροπολογίας 93. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 Βλάστο. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 96 Evans. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 95 Blockland. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 του εισηγητού ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 Ζαμπόφσκι 98 στόκμα ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 99 της 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 για Ζεμπόφσκι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 του συγκητή υπέρ κατά αποχές θα γίνει ηλεκτρονικός έλεγχος. Τέλος. 18 υπέρ, 15 κατά, εγκρίνεται 22 του συγγετή. 103 καλύπτεται, από την 22 πάμε Καταπίπτει και επόμενη, η Τζούρι 5. Πάμε στην 104 για Ζεμπόφσκι υπέρ. Κατά. Αποχές, απορρίπτεται. 23 του συγκητή υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος. 17 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται. 105 Evans, καταπίπτει. Falls 105 Evans. Ψηφίζουμε την Evans 105 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 106 για Ζεμπόφσκι. Ταυτόσημη με την Ζούρι 6 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 107 βλαστό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται της νομικής η 7 υπέρ η τζούρι 7 κατά αποχές απορρίπτεται τζούρι 8 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 Λίχτενμπέργκερ είναι ταυτόσιμη με το 109 Εύανς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβιβαστική C λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρθρο 18 παράγραφος 1, 110 τέλος πάντων του Κύρικο Πίπερ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 της νομικής υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 του φυγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 κυρκόπ πίπερ, κατά αποχές απορρίπτεται 10 της νομικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 113 για Ζεμπόσκι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 115 Στόκμαν καταπίπτει 114 καταπίπτει 117 Γένσεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 Κίρκοπ υπέρ κατά δεν ξέρω πρέπει να ελέγξουμε την 116 Κίρκοπ ξεκινάει πέρας 14 ψήφοι υπέρ 20 ψήφοι κατά απορρίπτεται λοιπόν η Κίρκοπ 11 της νομικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 κύρκοπ υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος 118 κύρκοπ Πέρας. 21 υπέρ, 12 κατά, εγκρίνεται. 119 γέννησεων υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 120 γέννησεων υπέρ. Αποχές εγκρίνεται. 25 της ηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 121 καταπίπτει. Δύο σε στο βιβασμό 27 του εισηγητού. 26 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκλίνεται, 122 Γένσεν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. 124 Κίρκοπ. ...124 λοιπόν υπέρ... ...κατά αποχές απορρίπτεται 123 Γένσεν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 125 κυρικό υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 12 αστυνομικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 αστυνομικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 για υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 128 συμπεριλαμβάνεται συμβαστική Συλλατινικό. λατινικό για Ζεμπόφσκι 127 το ίδιο Πάμε στην 133. Γιάννησεν. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 124 στόκμαν 134 στόκμαν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 135 δεγκράντες πασκουάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 136 μακάρθη και άλλοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 137 Λίχτενμπεργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 έχει καταπέσει 138 βλάστο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 ηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 του ηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 μακάρθη και άλλη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 15 της νομικής υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 140 μακάρτη και άλλη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 141 Evans υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στην 142 της ναι, υπέρ αποχές εγκρίνεται Βόρτμαν Κόλ 143 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 144 Βόρτμαν Κόλ κατά αποχές απορρίπτεται 145 Βόρτμαν Κόλ κατά νομίζω ότι απορρίπτεται θα κάνουμε επαλήθευση για την 145 Βόρτμαν Κόλ ψηφίσατε όλοι πέρασε 14 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 147 αντεγκάντ Πασκάλ υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 146 Πισκόρσκι υπέρ, κατά, δεν ξέρω, πρέπει να κάνουμε παλήθευση 146 Πισκόρσκι. Τέλος. 17 υπέρ, 17 κατά, δεν εγκρίνεται. 36 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 148 βόλτμαν Κόλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 149 Τεσσενέ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 150 Evans υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται πρέπει να κάνουμε παλήθευση για 150 Evans τέλος 17 υπέρ 15 κατά μια αποχή εγκρίνεται πίπτη 151 τεσσενέ τη λογική σκέψη 37 τεσσενέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 τεσσενέ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 Evans υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 40 είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2 τη ηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η πρώτη τροπολογία της νομικής υπέρ κατά εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη νομοθετική πρόταση. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Μάλιστα, τέλος ψηφοφορίας 21 υπέρ, 0 κατά, 13 αποχές. Ψηφίζουμε το νομοθετικό αυτό ψήφισμα, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 34 στις παρόντες 32 ψήφισαν, 18 υπέρ, καμία ψήφος κατά και 14 αποχές. Συγχαρητήρια στον κύριο Τέισενέ, τον εισηγητή. έκθεση Αλμπερτίνη για το δικαίωμα των επιβατών στα λεωφορεία και στα πούλμαν. Είμαστε έτοιμοι. Τοπολογία 41 Λίχτεμπεργκερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 42. Ζόμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 κάνουμε Πασκουάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 Μπράντμπορν και Κίρκοπ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται άρθρο 2 παράγραφος 2 τροπολογίας Ζαγεμπόση Γέγκελ Σόμερ είναι ταυτόσιμος υπέρ κατά Αποχές νομίζω ότι απορρίπτονται, αλλά ας κάνουμε μια επαλήθευση. Ξεκινά λοιπόν η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 34 παρόντες, 15 ψήφοι υπέρ, 19 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται λοιπόν η τρία του συγγητή υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα γίνει όμως ένας έλεγχος. Σας παρακαλώ. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 17 υπέρ, 16 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται η τροπολογία 3 του συγητή. Άρα καταπίπτει 46 τικάου, Πάμε στην 48, Grandes Πασκαλ, Σαν προστίκη υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 4 του συγκητή υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά ας γίνει ένας έλεγχος. Εγκρίνεται, μα τι λέτε. Το είπα και εγώ. Θέλω να το επιβεβαιώσω. Καμιά φορά ακόμα και οι καλύτεροι άνθρωποι που κάνουν προβλέψεις θέλουν κάποια επαλήθευση. Για να επαληθεύσουν και την ατότητα που έχει ο κ. Ζεμπόφσκι να προβλέπει και να διακρίνει τι γίνεται. Όπως είχε προβλεφθεί, έχουμε 23 υπέρ, 11 κατά, εγκρίνεται. 5 του συγγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 6 συγκριτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 51 μακάρτι και άλλοι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 κοχ είναι ταυτόσιμο με την Evans Τσικάου την 50 υπέρ κατά πολύ μικρή διαφορά θα κάνουμε παλήθευση Πέρας του ελέγχου. 15 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. 52 Φέρμπερ υπέρ. Κατά. Λοιπόν, και εδώ θα κάνουμε επαλήθευση γιατί είναι μπερδεμένα τα πράγματα. Ψηφίσατε όλοι. πέρας επαλήθευση, 17 υπέρ 16 κατά και καμία αποχή εγκρίνεται 52 Φέμπερ 53 Τεγκράν Πασκάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται Πάμε στην 54 Evans Tikau με την προφορική τροπολογία που γνωρίζετε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 55 Δεγκάν Πασκουάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 Bradford Kirkhope κατά αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας κάνουμε μια επαλήθευση για την Bradford 56 πέρασε επαλήθευσης 19 υπέρ 15 κατά εγκρίνεται Καταπίπτει η 57. Πάμε στην 58 Αλμπερτίνη. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 7 του εισηγητή. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 59 Αλμπερτίνη. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. Καταπίπτει η φουρέ η 60 και πάμε στην 61. Υπέρ. Κατά εγκρίνεται 62 Γέγκλ κατά αποχές εγκρίνεται 63 Γέγκλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 Γέγκλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 για σεμπόσκι Γέγκλ κατά αποχές απορρίπτεται 67 ευανστικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 66 τεγκράντς πασκουάλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 68 τεγκράντς πασκουάλ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 69, πάμε στην 70, δεν κάνει Πασκουάλ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 71 Φέρμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 72 Φέρμπερ υπέρ. Κατά. Αποχές νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε υπαλήθευση 72 Φέρμπερ. Τέλος. 15 υπέρ, 19 κατά, απορρίπτεται. Κοχ, 73 και 76 μαζί, υπέρ. Κατά. Όπως και πριν νομίζω. Λοιπόν, 8 του εισηγητή, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται, 74 γέγκλ υπέρ Κατά. Κύριο Σέβανς. Να ρωτήσω τι σημαίνει αυτό η 74. Δεν είναι σαφές. Είτε είναι αδύνατο, physically ή actually, στα αγγλικά δεν έχει διαφορά. Σωματικά δηλαδή, φυσικά ή πραγματικά. Εφόσον είναι δηλαδή αδύνατο, είναι αδόνατο. Δεν ξέρω, μπορεί σε κάποια άλλη γλώσσα να σημαίνει κάτι διαφορετικό αυτό που αναφέρεται, αλλά πραγματικά δεν βγάζει νόημα. Φυσικά, ο κ. Σεμπόφσκι φυσικά και έχει μεγάλη διαφορά. Εξαρτάται από τι γλωσσικέ σου ικανότητε, αγαπητέ Ρόμπερτ. Το ψηφίσαμε ήδη. Δεν έχει νόημα να κάτσουμε να ξανασυζητήσουμε αυτά που έχουμε ήδη ψηφίσει. Εκτός μικροφώνου τα σχόλια. Είναι πολύ απλό, Πρόεδρε, εφόσον από όσο ξέρω το ένα είναι αντικειμενικό και το άλλο είναι υποκειμενικό. Mm. Συνεχίστε. Mm. Θέλει ο ηγητής να παρέμβει. Όχι. Καλώς. Ψηφίζουμε την 74. Ε, τα, τα, μετά το συζητάμε το φιλοσοφικά το θέμα όσον αφορά το σημείο αυτό. Πρέπει να ψηφίσουμε την 74, υπέρ της 74. Κατά, αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η 9 του συγκητή, πάμε στην 75 για εγκλήπερ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 10 του συγκητή υπέρ, είναι ταυτόσιμο με την 77 για εγκλήπερ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 78 Evans Τσικάου υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 Φέρμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει ποια καταπίπτει καταπίπτει 80 πάμε στην 11 του συγκεκριτή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κατά πίπτη 81, πάμε στη 12 του εισηγητή που είναι με τον 82 κοχ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 83 Μακάρθη και άλλοι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έλεγχος, εντάξει. Ας ελέγξουμε λοιπόν την 83 Μακάρθη και άλλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 14 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. 13 του εισηγητή, ταυτόσιμη με το 84 κοχ υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 85 Εύαν Σικάο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 86 Αγιάλα Σέντερ, καλύπτεται από την 85, πάμε στο 87 κοχ, ταυτόσημη με την 88 Evans Τσικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 Μακάρτη και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 Evans Τσικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 14, 14 του συγκητή. 92 92 καταπίπτει και 93 και 90 και 94. Πάμε στη 15 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 96 Εύαν Τσικάου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 95 καταπίπτει. 16 του εισηγητή τώρα. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 98 Κοχ ταυτόση με την 99 Evans Τσικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 η άλλα σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 Κοχ ταυτόση με την 101 Evans Τσικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 102 κοχ ταυτόση με την 103 υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 105 Evans Τσικάο υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται 104 Γιάλα Σέντερ πίπτη 17 του συγητή τώρα που είναι ταυτόση με την 18 του συγητή. ψηφίζουμε μαζί τις δύο υπέρ κατά άποχες εγκρίνονται 106 Φέρμπερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 107 για Λεσέντερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 108 Ευαντσικάου υπέρ κατά επαλήθευση να κάνουμε έλεγχο. Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε έναν έλεγχο. 108 ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 16 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, μία αποχή εγκρίνεται. 109 για άλλα σέντερ υπέρ, κατά, Νομίζω ότι εγκρίνεται. Ας γίνει όμως επαλήθευση. Ξεκινάμε. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 9 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Άρα καταπίπτει 110. πάνω στην 111. ζώμερ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112. Bradburn Kirkhope υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 114. ζώμερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 115. Αλμπερτίνη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 113. Γέγκλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 του συγητή με προφορική τροπολογία που γνωρίζετε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 20 του συγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει έτσι η 116 Λίχτενμπέργκερ. Ναι, κατέπεσε. Πάμε στην 117 Αλμπερτίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 Αλμπερτίν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 119 Αλμπερτίν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 120 Αλμπερτίν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 121 Γιαζεμπόσκι Γέγκλ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 122 Αλμπερτίν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 123 Κοχ που είναι ταυτόση με την 124 Evans τη Kuiper Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 125 για Ζεμπόσκι Γέγκλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. 126 Γέγκλε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Συγχωρήστε με. Αλλά έχασα το μέτρημα. 126 υπέρ κατά δεν ξέρω έλεγχος επαλήθευση για την 126 γέγκλ τέλος 15 υπέρ 18 κατά απορρίπτεται 127 μακάρθη υπέρ κατά μου λείπουν χέρια επαλήθευση έλεγχος 127 Μακάρθη Μακάρθη και άλλοι 127 τέλος 18 υπέρ 13 κατά εγκρίνεται 128 κόχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πίπτη 21 του ηγετή 129 κόχ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 του ηγετή πίπτη 130 Evans κάου με προφορική τροπολογία που ξέρετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 131 καταπίπτει η Λίχτεμπεργκερ και πάμε στην 132 Γέγκλ που είναι ταυτόσιμη με 133 Φέρβερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 του συζητητή υπέρ, κατά, πρέπει να κάνουμε επαλήθευση όσον αφορά την 23. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 22 υπέρ, 11 κατά υπέρ. Σηκώνετε λίγο τα χέρια σας. Είσαστε κουρασμένοι κι εσείς αλλά κι εγώ. 24 του συγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 25 του εισηγητή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει 135 και 134 στην 136 πάμε. Μακάρθη και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 137 Evans κάω υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 του ηγετή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται πάμε στα παραρτήματα 138 Bradburn και Κίρκο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 139 Εύαν Τσικάου με προφορική τροπολογία που τη γνωρίζετε υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Αιτιολογικές σκέψεις 29 Αλμπερτίνη υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 30 Εύαν Τσικάου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 31 Αλμπερτίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 32 Σόμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 1 του εισηγητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ κατά Λιχτονικός έλεγχος για τη 36 Λίχτεμπεργκερ. ξεκινάμε Πέρας. 15 υπέρ, 18 κατά. Απορρίπτεται. 38 τώρα. Εύαν Στικάου. Ζητώ συγγνώμη. Ποιος είναι υπέρ, λέει ο πρόεδρος. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Καταπίπτει 37 κοχ, 2 του συγκητή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 Evans Τσικάου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 Γέγκλερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεχόμαστε και τις διάφορες μεταθέσεις Σόμερ, Λιχτεμπέργκερ κλπ. τετολική σκέψη 8 και κλπ. Ψηφίζουμε νομοθετική πρόταση που τροποποιήθηκε. Ξεκινάει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Λείπει μία ψήφος. Τέλος πάντων. Πέρας. 33 παρόντες, 32 ψηφίσαντες, 32 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή. Πολύ καλά λοιπόν για τον κύριο Αλμπερτίνη και στέφεται επιτυχία του ψηφίζοντας το νομοθετικό αυτό ψήφισμα που ξεκινάει αυτή τη στιγμή. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Λοιπόν, 33 ψήφοι πέρα αυτή τη φορά, 0 αποχές, 0 ψήφοι κατά. Allora, abbiate pazienza, Να έχετε υπομονή γιατί έχουμε και κάποια πραγματάκια να κάνουμε. Έχουμε μια εκθεσούλα που αφορά το συμπολίτη μου, τον Μάρκο Πόλο. Ψηφίζουμε την έκθεση λοιπόν όσον αφορά το πρόγραμμα Μάρκο Πόλο 2 τη χορήγηση οικονομικής βοήθειας, τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσης όσον αφορά το σύστημα μεταφοράς εμπορευμάτων. Κύριε Στόκμαν, εισηγητής μας. Ψηφίζουμε, παρακαλώ. Σας παρακαλώ Όσοι θέλετε να συνομιλήσετε παρακαλώ βγείτε από την αίθουσα. Ψηφίζουμε τη συμβαστική πρόταση. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές η συμβαστική πρόταση γίνεται δεκτή. Οπότε καταπίπτουν όσα καλύπτονται από αυτήν. Τροπολογία 12, Μπλόκλαντ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 13. Καταπίπτει. Ε, προφορική τροπολογία Στόκμαν, συγγνώμη. Τροπολογία 1 προφορική. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16. Βόρτμαν Κόλ με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτό. Τροπολογία 2 του εισηγητού με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. 17, Λίχτεμπεργκερ, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Στόκμα με προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 20 καταπίπτει. Το ίδιο και η 4, 18, 19, όλες αυτές έχουν καταπέσει. Τροπολογία Στόκμαν 5, προφορική, ποιος είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 6, Στόκμαν υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 7, Στόκμαν, Ποιο είναι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Προφορική τροπολογία 8 Στόκμαν. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 21 Λίχτεμπεργκερ. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 22 Λίχτεμπεργκερ. Υπέρ. Κατά αποχές. Εγκρίνεται. 23 Τσικάου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίπτεται. 24 Λίχτεμπεργκερ. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 Λιχτεμπέργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 Τσικάου ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 27 Στόκμαν με προφορική τροπολογία 9 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 Τσικάου ποιος είναι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 29 Στόκμαν με προφορική τροπολογία 10. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 30 Τσικάου. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 31 Στόκμαν με προφορική τροπολογία 11. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 Στόκμαν με προφορική τροπολογία 12. Υπέρ. Κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 32 Στόκμαν με την προφορική τροπολογία 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε. Τέλος ψηφοφορίας. Συγγνώμη. Σημερίζομαι την ευθύνη. Ε, δεν φταίτε εσεί δικό μου το λάθος. Μέα κούλπα, 32 εγκρίνεται, 33 τσικάω. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. προφορική τροπολογία 13 Στόκμαν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στόκμαν τροπολογία 14 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Βόρτμαν Κόλ 34 υπέρ. Κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά κάνουμε έναν έλεγχο. Πέρας. 19 υπέρ, 14 ψήφοι κατά. Εγκρίνεται η Βότμαν Κόλ 34 και έτσι καταπίπτει η 35 Μπλόκλαν. Πρέπει να ψηφίσουμε όμως 36 Μπλόκλαν υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Πάμε στην 6. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Του εισηγητού η 1 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Στόκμαν, προφορική τροπολογία 15 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 7 αποσύρεται. 8 καλύπτεται από τη συμβαστική. Ψηφίζουμε λοιπόν την πρόταση νομοθετικού περιεχομένου σε τροποποιήθη. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. 33 υπέρ 0 κατά. Ε, άλλο ένα σλάμ. Λοιπόν, να επαναλάβουμε λοιπόν τα ίδια και στην, ε, στο ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ψηφίζουμε. Πέρας. 33 υπέρ, 0 κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια στον κύριο Στόχμαν, λοιπόν. Ορίστε. Ορίστε. Ήδη είχαμε 5 λεπτά. Και άλλα 5 λεπτά. Άλλα 5 λεπτά. Καλώς.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 May I ask all colleagues take the... Παρακαλώ συνάδελφοι καθίστε. For the final part of this long... vote... Για το τελικό τμήμα αυτής της μακράς ψηφοφορίας. Okay. Draft report the proposal of European... Πρόταση οδηγία Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου που καθορίζει το πλαίσιο για το μεταφορικό σύστημα στο το τομέα των δικών μεταφορών και διαπαφέ με άλλου τρόπου μεταφορά. Ευφυή συστήματα μεταφορών. Η κυρία Άννα Γένσεν είναι η συγγήτρια που ζήτησε το λόγο και τη τον δίνουμε. Well, Σα ευχαριστώ. Λίγε παρατηρήσει να κάνω μόνο. Η ψηφοφορία για την τροπολογία 45 Συμφώνησα με την κυρία Πατάκη που την υπέβαλε την τροπολογία να ενταχθεί στο άρθρο 4 και όχι στο άρθρο 3α νέο. Για την ψηφοφορία 58 του κυρίου Σαβαρή θα ήθελα να ψηφιστεί ως προσθήκη. Και τέλος, να πω ότι οι σοσιαλιστές επίσης συμφωνούν με τους εμβιβασμούς 3 και 4, άρα έχουμε κατά πάσα πιθανότητα πλειοψηφία. Benissimo. Ωραιότατα. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την ψηφοφορία μας. Πριν ξεκινήσουμε, έχω τη χαρά να γνωστοποιήσω στους συναδέλφους ότι έχουμε εκπροσώπους της Γερμανικής Βουλής, της Bundestag, που και οι συνάδελφοι ευτυχώ ή δυστυχώ ασχολούνται με τις μεταφορές και είναι εδώ μαζί μας σήμερα. Καλώς ήρθατε όλοι σας. Λοιπόν, ψηφίζουμε την τροπολογία 25 Σαβαρή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 26. Κούστασερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 33. Κούστασερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 2 του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 1 υπέρ. Σε δύο τμήματα ξεχωριστά πρώτο τμήμα υπέρ του πρώτου τμήματος. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και το δεύτερο τμήμα. κατά πίπτη 35 ή 36 ή 34 ή 3 της ηγήτριας Παραμένει όμως η 37 Γένσεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 και αυτή κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν οι 41, 40, 38, 39, 2 τις εισηγήτες λέει ο, ο Προεδρός, οι 4 μάλλον εννοεί και πάμε 42 Σαβάρι υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 5 εισηγήτριας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν οι 44, οι 6. Πάμε στη 43, υπέρ, κατά. Νομίζω ότι εγκρίνεται, ας κάνουμε μια επαλήθευση. 43, μπάρση πατάκι ηλεκτρονικός έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. 19 υπέρ, 14 κατά, εγκρίνεται λοιπόν η τροπολογία. 46 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 εισηγήτριες υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 της ηγετρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 50 τσικάο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 ράκ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 της ηγετρίας υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 52 Παναγιωτοπούλου Κασιώτου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 45 Μπάρση Πατάκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 10 της υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 53 Σαβαρή υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά κάνουμε μια παλήθευση πέρας 14 υπέρ 17 κατά καμία αποχή απορρίπτεται 54 μπάση πατάκι υπέρ κατά Νομίζω ότι εγκρίνεται. 11 της υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 Γέντσεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 56 Γέντσεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 Γέντσεν υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 12 εισηγήτρες υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 με προφορική τροπολογία που ξέρετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 Γένσεν προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 Σαβαρή κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 62 γένσεν, κάποιες διορθώσεις υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 13 εισηγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 14 της εισηγήτριας υπέρ, κατά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 Γένσεν υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 73 βάση πατάκι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 72 κατά τμήματα φουρέ. Πρώτο, η πρώτη προπαράγραφος υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα, κατά πίπτη. Πάμε στην 20 συγγήτριας υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 21 εισηγήτριες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 μπάρση παθάκι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 γένσεν με προφορική τροπολογία που ξέρετε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 προστασία δεδομένων συγγνώμη Λάχτριντ υπέρ κατά επαλήθευση έναρξης αυτής 16 υπέρ, 18 κατά, απορρίπτεται. 78 λάχτρια υπέρ, κατά. Νομίζω ότι είναι τα ίδια όπως πριν. Απορρίπτεται 79 Τσικάο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται 80 Ρακ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 μπάση και υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτουν 82 κούστας 22 εισηγήτριας. Αποσύρεται 23. Πάμε στην 24 της εισηγήτριας. Υπέρ. Κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 27. Γένσεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 28. Αποσύρεται. 29. Γένσεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 30. Γένσεν υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31. Τσικάου υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 1. Εισηγήτριας υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. δηλαδή. Ρακ υπέρ κατά άποχες εγκρίνεται. Ψηφίζουμε την τροποποιημένη νομοθετική πρόταση και ξεκινάμε. Ψήφισατε όλοι. Πέρας. 35 παρόντες 34 ψηφίσατε, 32 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Ψηφίζουμε το ψήφισμα νομοθετικού περιεχομένου. Ξεκινάμε. Πέρας. Όπως πριν, 32 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή. Πολλά συγχαρητήρια στην κυρία Γένσεν. και ελπίζουμε να επαναληφθεί αυτό σε μερικά δευτερόλεπτα, διότι έχουμε την έκθεση πρωτοβουλίε όσον αφορά τα ευφυή e συστήματα μεταφορών και το σχέδιο δράση που το ανέλαβε η κυρία Γένσεν. Τροπολογία 1. Κούστα Σερ. Δεν είναι αποδεκτή αυτή. Τροπολογία 3. Μπάρση Πατάκη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Επιτροπή Περιφερειακής Πολιτικής Τροπολογία Άννα υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Εγκρίθηκε. Να κάνουμε επαλήθευση για να δούμε αν εγκρίθηκε. Πέρας. Βέβαια με μεγάλη διαφορά εγκρίθηκε. Όπως έλεγε ο κύριος Γιαζεμπόφσκι Πρέπει να είστε προσεκτικοί, ε. Ρέτζι 2 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 4 ακούστε σε υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση πρέπει να γίνει. Πέρας. 14 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. Ζρέτζι 3 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5 κούστασορ υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 6 μπάση πατάκι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 7 μπαρσιπατάκι πατάκι υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 8 μπαρσιπατάκι πατάκι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 9 μπαρσιπατάκι πατάκι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 κούστα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11 Λάιχθριτ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 12 τσικάου. Κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ε, ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 φουρέ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 φουρέ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 15 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 16 Σαβαρή. Έλεγχος. Καλός. Επαλήθευση για 15 Μαρινέσκου. Πέρας. Πολύ σωστό. Έκανα λάθος εγώ. Εγκρίνεται. 28-7. 16 Σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 17 σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 σε 20-2σαρίπερ. κατά Αποχές. Απορρίπτεται. 21 Μαρινέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 22 Μπάση Πατάκη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 23 Μαρινέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 24 Μαρινέσκου. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 25-24 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 26 Κούστας κατά νομίζω ότι εγκρίνεται 27 Κούστας έλεγχος να δούμε αν εγκρίνεται 26 λοιπόν Ναι, ψήφισα λάθος. Γι' αυτό ερμήνευσα και τα αποτελέσματα λάθος. Πέρας ψηφοφορίας. 14 ψήφοι υπέρ, 20 ψήφοι κατά, απορρίπτεται 27 κουστάσερ υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται 28 τσικάο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται 29 λάχτφριντ υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται. 30 τικάο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31 κούστασερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 32 τσικάο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 33 κούστασερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 8 υπέρ 8 συγγνώμη κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Κούστασερ 2 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Αιτιολογική σκέψη ε, αρχικό κείμενο με προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τελική ψηφοφορία που ξεκινάει. 36 παρόντες πέρας ψηφοφορίας ψηφίσατε 36, 34 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, καμία αποχή. Ξανά συγχαρητήρια προς την κυρία Γένσεν. Ανανεώνουμε τα συγχαρητήριά μας. Λοιπόν, πάμε στη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Πακιστάν υπέρ κατά πρέπει να ξεκινήσουμε, να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ξεκινάει η ψηφοφόρια. Πέρας. 36 ψηφίσατε, 36 υπέρ, καμία ψήφος κατά, καμία αποχή, όλα εντάξει. Όμως, ο, πρόταση του Συμβουλίου Απόφασης για το πρωτόκολλο της εφαρμογής για τα συστήματα ή το μεταφορικό πρωτόκολλο για την περιοχή των Άλπαιων, τη σύμβαση των Άλπαιων. Σχέση εκθέσεως για την πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου για τη σύναψη τη σύμβαση των Άλπαιων στον τομέα των μεταφορών. Ψηφίσατε όλοι. Ωραία. Τέλος ψηφοφορίας. 36, 0, 0. 36 υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Πράσινη βίβλος για το μέλλον της πολιτικής δομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Μισό λεπτάκι, διότι μετά αυτή τη ψηφοφορία, την τελευταία ψηφοφορία, α, υπάρχει και άλλη μετά. Μετά τις δύο ψηφοφορίες, ο καθένας από εσά έχει ανηλυμένες υποχρεώσεις και αυτή είναι η τελευταία μας συνεδρίαση και ε, θέλω να πω δύο λόγια από την πλευρά μου, μόνο δύο λόγια. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά εκ βάθους καρδίας όλους σας για τη δουλειά που κάναμε μαζί, που ήταν υπέροχη δουλειά δουλειά που κατά ε, την άποψή μου επέτρεψε στην Επιτροπή μας και αυτές οι ψηφοφορίες το δείχνουν και 36.00 θυμάμαι και 46.00 όλες αυτές οι ψηφοφορίες δείχνουν ότι εκφράζουμε αλληλεγγύη και συμβάλαμε πραγματικά στην ευρωπαϊκή πολιτική. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν συμμερίζεστε εσείς τη δική μου άποψη αλλά πώς να το πω ότι το φλάμπουρο ή η δάδα της Ευρώπης ε, βγαίνει από το κοινοβούλιο περισσότερο από ότι από τα θεσμικά όργανα. Το Συμβούλιο κάνει διακυβερνητική δουλειά εξορισμού. Πρέπει να πω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ειλικρινά κατά την άποψή μου εκφράζει κάπως αδύναμα τη δυνατότητα που έχει να εκφράζει την Ευρώπη. Σίγουρα το Κοινοβούλιο το κάνει αυτό με πολύ καλύτερο τρόπο κατά την άποψή μου και αυτή η Επιτροπή είναι η Επιτροπή που πάει καλύτερα από τις άλλες. Καταφέρνει πάντα να βρίσκει τις σωστές ισορροπίες, ούτως ώστε να υπάρχει η Ευρώπη, να συμβάλλει θετικά σε αυτά που γίνονται η Ευρώπη. Ε, λοιπόν και αναγνωριζόμαστε και εκτός αυτής της αίθουσας και εκτός των θεσμικών οργάνων αυτά που κάνουμε. Συνοψίζοντας όλα αυτά πρέπει να πω ότι αυτή είναι η μοίρα συχνά εκείνων που κινούνται πολύ καλά και δεν αναγνωρίζονται οι προσπάθειες επαρκώς. μπορούμε να αυτοσυγχαρούμε, να συγχαρούμε τους αυτούς μας, να είμαστε ευχαριστημένοι αυτά που κάναμε. Είμαι σίγουρος ότι οποιοδήποτε επιστρέψει στην επόμενη πενταετία θα συνεχίσει αυτή τη δουλειά που ξεκινήσαμε αυτά τα χρόνια για τα αποτελέσματα που πετύχαμε ήταν θετικότατα. Για να τα κλείσουμε αυτά, ετοιμάσαμε μικρή έκπληξη, ένα μικρό δώρο. Και τι είναι, χάρη, για μια ακόμη φορά στη δουλειά, την πολύ αποτελεσματική, αποδοτική δουλειά της κυρίας Κάσνιτς και όλης της γραμματείας που πραγματικά μας βοήθησε η γραμματεία, μπορώ να το πω αυτό, μας βοήθησε με υπέροχο τρόπο στις δουλειές μας, θέλαμε να μαζέψουμε όλα τα briefing notes και όλες τις εκθέσεις που ετοιμάσαμε. Ένα μικρό βιβλιαράκι ετοιμάσαμε, ένα φάκελο όπου έχουμε ολόκληρη την ιστορία των, ε, της πενταετίας μας, και μπορώ να προσθέσω και μία μικρή εισαγωγή που λέει αυτά τα πράγματα που είπα τώρα. Ο καθένας από εμά θα είχε αυτό το βιβλιαράκι. Άντε σε ένα μήνα το πολύ και πιο πριν ίσως να τυπωθεί αυτό το βιβλιαράκι που ε, με τακτικό τρόπο θα συνοψίζει όλα αυτά που κάναμε. Θα δείτε από αυτή την άποψη ποια είναι τα μικρά συνεχή βήματα που κάναμε εμείς, που προξενήσαμε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα βήματα που κάναμε να κάνει η μεταφορά, να το μέσο των μεταφορών. Ευχαριστώ όλους και συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Όπως πάντα, την τελευταία λέξη την έχει και ο Ζιαζεμπόφσκι. Λίχτεμπεργκερ. Κύριε Λίχτεμπεργκερ. Να κάνουμε και μια δεύτερη ψηφοφορία για, την, ε, για το παλαιό πρωτόκολλο μεταφορών, γιατί ψηφίσαμε μόνο... Δεν ψηφίσαμε ακόμα μόνο το νομοθετικό ψήφισμα. Ψηφίσαμε μία φορά μόνο, Πρόεδρε. Nice ε, Καλώ. Καλώς. Τα συναισθήματα μας, κάνει να κάνουμε, μας κάνουν να κάνουμε λάθη λοιπόν. Λοιπόν, διορθώσουμε το σφάλμα, ξεκινάει η ψηφοφορία. Ωραιότατα ψηφίσατε όλοι, μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Πέρας. 35-0-0 όλα μια χαρά. Ρυθμίσαμε και τις Άλπεις, τις βολέψαμε. Λοιπόν, έκθεση πρωτοβουλίας όσον αφορά την πράσινη βίβλο για το μέλλον τη πολιτική στον τομέα των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών. Η κυρία Εύα Λίχτεμπεργκερ, συγγήτρια, ψηφίζουμε τροπολογία 1. Λίχτεμπεργκερ, υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Τροπολογία 2, Λίχτεμπεργκερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3, Αγιάλα Σέντερ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 4, Σαβαρή. Υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Κάνουμε παλήθευση όμω, Ξεκινάμε. Τέλος. 15 υπέρ, 20 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται 5 σαβαρή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 6 σαβαρή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 σαβαρή υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 8 σαβαρή υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 για άλλα σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 Λίχτενμπέργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 10 Grand Pascal υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 12 Γέγκλε Φέρμπερ και 13 Βένετο Αλμπερτίνη ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε και τις δύο υπέρ. Κατά νομίζω ότι εγκρίνονται. Έλεγχος, έλεγχος. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. 20 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Συμβαστική α. Καταπίπτει. Δεκαεπτά τσικάω υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 18 τσικάου κατά τμήματα πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται δεύτερο τμήμα κατά πίπτη αυτό 19 Βένετο Αλμπερτίνη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 Αγιάλα Σέντερ σαν προστίκη υπέρ κατά Πρέπει να εγκρίνεται, αλλά κάνουμε μια επαλήθευση. Ξεκινήσαμε τώρα. Ξεκινάει. Πέρας. 17 υπέρ, 18 κατά, καμία αποχή. Δεν εγκρίνεται. 21 gun. Χάττον υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται όχι επαλήθευση λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος πέρας 17 υπέρ 18 κατά δεν εγκρίνεται 22 κατά τμήματα Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 23 Φερνάντες. Σαν προστίκη. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. 24 Καταπίπτει 25 σαβαρή υπέρ. Κατά. Άποχες. Έλεγχος. Πέρας. 22 υπέρ, 13 ψήφοι κατά, εγκρίνεται. 26 Σαβαρή υπέρ, κατά, άποχες. Είναι κάπως αβέβαια τα χέρια σας, ε, παιδιά. Μπορούμε να ξαναδοκιμάσω σας παρακαλώ. 26 Σαβαρή υπέρ, κατά, άποχες, εγκρίνεται. 26 έλεγχος. Πέρας. Δίκαιο έχετε 15 υπέρ 20 κατά. Απορρίπτεται 27 σαβαρή υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική β υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει έτσι η Ζόμερ 28, η Μαρινάσκου 29, η 30, 31, 32, 33, 34, 35 και φτάνουμε στην 36. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά νομίζω ότι εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα έλεγχος ρώτοντα επαλήθευση λοιπόν όσον αφορά το δεύτερο τμήμα πέρας 20 υπέρ 15 κατά καμία απόχη εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα 37 τσικάω κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα. κατά πίπτη. 38 Αγιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά κάνουμε παλήθευση. Τέλος. 15 υπέρ 19 κατά. Καμία αποχή απορρίπτεται. 39 Στόκμαν κατέπεσε λόγω συμβαστική. 40 free υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 41 free υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται 42 λάχθροι δίπερ Κατά. Αποχές απορρίπτεται 43 λάχθροι δίπερ Κατά. Αποχές απορρίπτεται 44 Watman Call Κατά. Αποχές Νομίζω ότι εγκρίνεται. 45 Γέγκλε Φέρμπερ. Καταπίπτει λόγω της 44. 46 λοιπόν Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 47 ή 48. 49 τώρα. Λάιχτφριντ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική C λατινικό. Ποιος είναι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει λοιπόν η 50. Πάμε στην 51 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 55 Λίχτεμπεργκερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 53 ρακ σαν προστίκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 54 χάουτον σαν προστίκη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 57 Παναγιωτοπούλου Κασιώτου είχε προσερθεί 58 Λίχτεμπεργκερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 60 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική δι λατινικό υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν 61 62, 63 Παναγιωτοπούλου Κασιώτου, 64 Μαρινέσκου και 65. 66 Βόρτμαν Κόλ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 68 Γέγκλε Φέρμπερ με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 69 Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 70 αλλά υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ας γίνει μια επαλήθευση Πέρας. 15 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται 71 γέντσαν υπέρ. 71 ένα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 72 Γένσεν υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση. Πέρας. 13 υπέρ, 19 κατά, καμία αποχή. Απορρίπτεται. 73 Γένσεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 76 Αγιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 75 Γένσεν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 74 ρακ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 77 σαβαρή υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 78 γέγκλε φέρμπερ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται απορρίπτεται καλώς 79 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 80 Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ κατά άποχες νομίζω ότι εγκρίνεται αλλά ας γίνει μια παλίδευση. Chiusa la Πέρασε επαλήθευσης. 19 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβαστική ε υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 81, 82 και 83. 84 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά. Αποχές δεν ξέρω, επαλήθευση. 84 Μαρινέσκου. Πέρας. 19 υπέρ, 15 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται 85 κόστα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 Παναγιωτοπούλου Κασιώτο Πεσίρθη 87 Χάουτον υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 88 Μαρινέσκου υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 89 Τσικάου υπέρ κατά αποχές επαλήθευση Πέρας. 15 υπέρ, 19 κατά. Απορρίπτεται. Συμβαστική F υπέρ. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Κατά. Νομίζω ότι υπορρίπτεται, αλλά πρέπει να κάνουμε επαλήθευση. Άντε, δύναμη. Επαλήθευση για την συμβαστική εφλατινικό. Πέρας. Μάλιστα, δεν εγκρίνεται. 15 υπέρ, 18 κατά, καμία αποχή. Ψηφίζουμε την 90. Αγιάλα Σέντερ, λοιπόν, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 91. Λάιφτριντ, υπέρ. Η 90 κάνει να καταπέσει 91, η 92, η 93, και 94. Πάμε στην 95. Γέγκλε Φέρμπερ. Υπέρ. Κατά επαλήθευση. Ξεκινάει για την 95. Τέλος. 17 υπέρ, 17 κατά, καμία αποχή δεν εγκρίνεται. 96 Μαρινέσκου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 97 Τσικάου υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 98 Λάιχτ Φρίντ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 99 Κώστα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 100 σαβαρή κατά τμήματα, πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 101 σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 102 σαβαρή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 103 Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 104 Καταπίπτη, όπως και 105 και 106 107 τώρα Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 108 Βένετο Αλμπερτίνη. Ταυτόση με την 110 Κώστα Στέρξ υπέρ. Κάτα αποχές εγκρίνεται. 109 Γκριγκάν Πασκουάλ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 111 Κώστα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 112 Μπέργκερ υπέρ. Κατά Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 1 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 2 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 3 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 4 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 5 υπέρ. κατά αποχές εγκρίνεται Ρέτζι 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ρέτζι 7 υπέρ κατά έλεγχος για τη Ρέτζι 7 Τέλος. 11 υπέρ, 23 ψήφοι κατά. Απορρίπτεται μεγάλη πλειοψηφία. Ρέτζι 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ρέτζι 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ρέτζι 10 υπέρ. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 11 υπέρ. Κατά. Δεν ξέρουμε. Επαλήθευση. Πέρας. 11 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά, δίκαιο έχετε. Λοιπόν, η 12 καταπίπτει, Ρέτζι 13. Υπέρ. Η Ρέτζι 12 καταπίπτει. Ρέτζι 13 ζει ακόμα. Εκτός αν τη σκοτώσετε τώρα. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Σκοτώθηκε. Πάει. Ρέτζι 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Τέρμα. Ρέτζι 15 υπέρ. Κατά αποχές και αυτή τέρμα. Τελική ψηφοφορία που ξεκινάει. για το, τροποποιημένο, για το τροποποιημένο ψήφισμα. Τέσσερις υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Ευχαριστούμε και όλους μας και τον κύριο Λίχτεμπεργκερ, για την κυρία Λίχτεμπεργκερ μάλλον, για την έξοχη δουλειά της. Θάρρος, κουράγιο. Φτάσαμε στο σχέδιο δράσης για την αστική κινητικότητα. Σταρ ο κύριος Ζιλ Σαβαρή, πρωταγωνιστή. Λοιπόν, 14α νέα, τροπολογία 1, κράμερ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτουν οι 12 και οι 13 Πάμε στην, στην τροπολογία εισηγητή, προφορική τροπολογία για το ΣΥΒΙΤΑΣ. Λοιπόν, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αγιάλα Σέντερ, προφορική τροπολογία 14 υπέρ. Κατά. Νομίζω ότι απορρίπτεται, όμως πρέπει να κάνουμε παλήθευση. Αγιάλα Σέντερ, με προφορική τροπολογία 14. Τέλος. 16 υπέρ, 16 κατά. Καμία αποχή. Δεν εγκρίνεται. 15 Higgins υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 16 Σαβαρή Ρακ και λυπή, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 Σαβαρή Ρακ και λοιπά υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 18, 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 20 Ζόμερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 Κράμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 22 χίγγινς υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 χίγγινς υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 Σαβαρή Ρακ και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 σαβαρή κ.λπ. και λοιπά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Blockland προφορική τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 28 29 Αγιάλα Σέντερ υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται. 30. Μποπούι Πισκόρσκι υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 31. Σαβαρή Ρά κλπ. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32. Τσικάου υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται λέει ο πρόεδρος. 33. Ζόμερ υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 34 κράμερ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία του εισηγητή υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει αντα, 35 χάτων υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 σόμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 μποπούι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 μποπούι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 σαβαρή κλπ υπέρ τα αποχές εγκρίνεται 40 σόμερ υπέρ κατά άποχες Μ, απορρίπτεται 41 τσίκα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 42 ζόμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 43 σαβαρή και υπόλοιποι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 44 Kramer υπέρ. Δίκιο έχετε. Καταπίπτει. Η 45 Σαβαρή και άλλοι υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 Kramer υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτε 47 για Λασέντερ υπέρ Κατά αποχές απορρίπτεται 48 Kramer υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 49 χάτων υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 50 τσικάου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 51 τσικάου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 52 τσικάου υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 53 ζόμερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 Σαβαρή Ρακ και άλλοι κατά αποχές εγκρίνεται καταπίπτει 55 Ψηφίζουμε το δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται το δεύτερο τμήμα 56 Γιάλα Σέντερ καταπίπτει όχι α δεν καταπίπτει μάλιστα «56 Γιάλα Σέντερ υπέρ» κατά απορρίπτεται «57 Γιάγκλε Φέρμπερ» κατά αποχές απορρίπτεται 58 ζόμερ ταυτόσημη με την 59 υπέρ κατά απορρίπτεται 60 γέλα σέντερ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 61 Βόρτμαν Κόλ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 Ζόμερ ταυτόσημη με την 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 64 βαρύ και άλλοι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 χώτων υπέρ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 66 Αγιάλα Σέντερ υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 67 Παναγιωτοπούλη υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. 68 Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 69 Γέγκλε Φέρμπερ υπέρ. Κατά απόχέ απορρίπτεται. 70 Σαβαρή και λοιποί υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δύο ζώμερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τρία κρέμερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Τέσσερα γέγκλε φέρμπερ υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Πέντε ζώμερ υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 6 ζώμερ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 7 ζώμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 8 χάτων υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 9 βατάνεν υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 10 ζωμερ υπέρ. Αποχές εγκρίνεται 11 ζωμερ υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ρέτζι 1. Α, όχι, καλύπτεται την λογική σκέψη ή λατινικό. Καλός παράγραφος 2, Ρέτζι, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 3, Ρέτζι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Παράγραφος 4, Ρέτζι, κατά τμήματα, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, δεν ξέρουμε, πρέπει να κάνουμε παλήθευση για το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 4 Ρέτζι. Ξεκινάει ο ηλεκτρονικός έλεγχος, το δεύτερο τμήμα της παραγράφου 4 Ρέτζι, που αφορά και προωθεί τον τουρισμό, εν προμό tourism. Λοιπόν, 10 υπέρ, 21 ψήφι κατά, απορρίπτεται, παράγραφος 5 Ρέτζι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, παράγραφος 6 Ρέτζι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 7 ρέτζιπερ κατά αποχές εγκρίνεται παράγραφος 8 ρέτζιπερ κατά αποχές απορρίπτεται τελική ψηφοφορία που ξεκινάει τώρα όσον αφορά το τροποποιημένο ψήφισμα Τέλος. 28 υπέρ, μία ψήφος κατά, δύο αποχές και αυτό το ψήφισμα πάει και με αυτό τελειώσαμε την ψηφοφορία μας. Ορίστε. Θα ήθελα να προτείνω να κοιτάξουμε το θέμα για τα σλότ ε. σήμερα το απόγευμα. Δεν έχουμε χρόνο να το συζητήσουμε πλέον σήμερα το πρωί. Σε πέντε λεπτά τώρα δεν προλάβουμε. Λυπάμαι. Εγώ θα ξανάρθω, ναι, θα ξανάρθω. Όλοι όσοι ενδιαφέρονται θα επανέλθουν.